ο Υπουργός ε, Αλεξάνδρ Βάντρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Σε αυτή την προχωρημένη ώρα θα αναφερθώ στι θέση του Συμβουλίου αναφορικά με το κέρας Αφρικής. Το κέρας της Αφρικής ε, αποτελεί μια περιοχή η οποία αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση και προκαλεί επίσης και διάφορες εντάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και είναι έτοιμη να αναμειχθεί έτσι Γνωρίζω πως το Ευρωκοινοβούλιο ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις. Η επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε η ελπισοπία σας το 2008 στην Ερυθρέα και την Αιθιοπία, αλλά και στο Τζιμπουτί. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Επίσης έχω καταγράψει τα ψηφίσματα για το κέρας Αφρικής, τα οποία έχετε επεξεργαστεί μετά από την επίσκεψη στην περιοχή. Θα πρέπει να αναφερθούμε στην σημασία που έχει το κέρας Αφρικής για την Ευρώπη. Από πλευρά Συμβουλίου καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλει το Κοινοβούλιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν προκλήσεις στην περιοχή. Υπάρχουν διάφορες πηγές έντασης ε, στο κέρας Αφρικής και θα αναφερθώ αργότερα σε λεπτομέρειες. Πάντως, κατά άποψη του Συμβουλίου αυτές οι εντάσεις ε, συνδέονται με τις εξελίξεις στην περιοχή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Συμβούλιο προσπαθεί να ενημερωθεί όσο είναι καλύτερο για τις εξελίξεις και τις συγκρούσεις στην περιοχή. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν αυτών των ε, διενέξεων των σειράξεων στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια διαφορά με την Αιθιοπία και την Ερυθρέα η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια από τις βασικές αιτίες της αστάθειας που επικρατεί στην περιοχή. Και αυτό αντανακλάται στα εξής. Υπάρχουν ε, ε, διάφορες ε, εμπόλεμες δυνάμεις στην περιοχή και υπάρχουν επίσης και πολλές ομάδες εμπολέμων και πολεμαρχών στην Αιθιοπία. Η Ερυθρέα έχει αποχωρήσει από τον AGFD και τέλος, οι σειράξεις στην Σομαλία έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική τραγωδία. Μία από τις σημαντικότερες που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο σήμερα. Τώρα, οι δραστηριότητε των πειρατών στις ακτές Σομαλίας είναι επίσης μια άλλη σημαντική συνέπεια αυτής τωρα η δραστηριότητα των διαφορών. Ένα άλλο ζήτημα αφορά τον ε, ανταγωνισμό για πόρους ε, όπως ε, το είδωρ. Αυτό αυξάνει έντι περαιτέρω τις ε, συγκρούσεις ε, ανάμεσα σε φυλές και σε εθνοτικές ομάδες. Επίσης αυξάνει την ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, κάτι το οποίο συνεισφέρει στην μετανάστευση. Παράλληλα υπάρχουν και πολλές αλληλεξαρτήσεις περιφερειακού χαρακτήρα. αναφερθώ σε μερικέ αυτέ. Υπάρχουν ε, οι διαφορέ συνοριακέ. Οι ε, διαφορέ ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα, το Σουδάν και την Αιθιοπία, το Τζιμπούτι και την Ερυθρέα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν ως πηγή αστάθειας ε, στην περιοχή. Να τονίσω πως η βελτιωμένη περιφερειακή συνεργασία θα μπορούσε να καταλαγιάσει τις εντάσεις που προκαλούνται η διατροφική ασφάλεια είναι ένα άλλο θέμα σημαντικό. Η ανομβρία και η ξηρασία αλλά και οι πολλές πλημμύρες οδηγούν σε ένταση αυτών των διαφορών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το Νταρφούρ στη Σομαλία, αλλά και άλλες περιοχές του κέρατος της Αφρικής. Δεν είμαι βέβαιος ε, ότι αναφέρθηκα εξαντλητικά σε όλα τα προβλήματα, αλλά θεωρώ πως το ζήτημα αυτό χρειάζεται να επιληθεί σε κάθε μία από τις χώρες μέσα στο περιφερειακό πλαίσιο με τρόπο δίκαιο και διαφάνεια. Η πειρατεία αρχικά αφορούσε ένα μικρό τμήμα των ακτών της Ομαλίας. Όπως ε, γνωρίζετε εσείς μέλη του Κοινοβουλίου, οι δραστηριότητες των πειρατών αναπτύχθηκαν σημαντικά και τώρα απειλούν ακόμα και την ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και την ίδια την ασφάλεια της ναυσιπλοεία στον κόλπο του ΕΔΕΝ και στι ακτέ τη Τανζανία και τη Κένια. Υπάρχουν και κάποιε άλλες ελληνεξαρτήσει που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρώπη και στις χώρες του κέρδου Αφρικής και αναφέρομαι στην τρομοκρατία αλλά και στη μετανάστευση. Ποιες είναι λοιπόν οι δράσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει. Το βασικότερο πολιτικό μέσο το οποίο διαθέτει το Συμβούλιο, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ σήμερα, είναι ο πολιτικός διάλογος όχι μόνο με τις επιμέρους χώρες, αλλά και με τους εμπλεκόμενους στην περιοχή όπως η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη, η Σύνδεσμος των Αραβικών κρατών αλλά και η Κίνα. Πολιτικός διάλογος λοιπόν αποτελεί μια αμοιβαία δέσμευση στο πλαίσιο των συμφωνίων που έχουμε συνάψει με κάθε μια από τις χώρες της περιοχής. Ωστόσο ο διάλογος ε, γίνεται σε επίπεδο επικεφαλής των ε, κοινοτικών αποστελών και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε άμεση επαφή με τις αρχές των εμπλεκομένων χωρών και αποτελεί την ευκαιρία στο να ακούσουμε τις απόψεις τους αλλά και να εξηγήσουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι αντιλήψεις μας, οι ανησυχίες μας ε, επί κάποιων ζητημάτων. Συζητάμε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και θέματα των δικαιωμάτων. Επιπλέον, το Συμβούλιο διαθέτει και το μέσο της ε, πολιτικής ε, ασφάλειας ε, από το 2008, το Δεκέμβριο, το Συμβούλιο είχε αναπτύξει αυτό το μέσο προκειμένου να καταπολεμήσει την πειρατεία στις ακτές Σομαλίας. Πρώτον, μέσω του πυρήνα συντονισμού βασίζεται στις Βρυξέλλες και από το καλοκαίρι του 2008 η από το φθηνό του 2008 μέσω της ε, οργάνωσης ε, Αταλάντη. Θα αφήσω την Επίτροπο Φεροβάλνερ να μιλήσει αναλυτικότερα επί του θέματος διότι είναι εν μέρη υπεύθυνη. Φυσικά το Συμβούλιο προσπαθεί να καταστήσει πιο σαφή, πιο διάκριτη την ε, παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις ε, χώρες αυτές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να δώσω το λόγο στην κυρία Φερέρο Βάλνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Υφυπουργέ, αγαπητέ Σάσα, αγαπητά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια απέθυνε έκκληση για μεγαλύτερη προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάσταση στο κέρας της Αφρικής και σήμερα στη συζήτηση αυτή εδώ αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου Λουί Μισελ ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί αλλά ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον εκπροσωπώ. όχι μόνο επειδή το θέμα είναι τόσο σημαντικό αλλά και επειδή επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, χρειάζεται να κινητοποιήσουμε το ναυτικό μα για να καταπολεμήσουμε την πειρατεία. Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία τη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Επιτροπή και στη συνέχεια κατάρτισε σχετική έκθεση. Η εσωτερική κατάσταση στις χώρες του κέρατος δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αν δεν την ε, θεωρήσουμε σε αλληλεξάρτηση με την ε, γενικότερη κατάσταση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, προσέγγιση επιμένοντας σε θέματα πολιτικής και οικονομίας, αν θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα και να διατηρηθούν τα βασικά στοιχεία του κοτονού και να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Να δω τώρα τι γίνεται αναχώρα, να δούμε τι γίνεται αναχώρα, πρωτού καταλήξουμε σε μια γενική στρατηγική. Καταρχάς να πω δύο λόγια για την Αθιοπία και την Ερυθρέα, κύριε Πρόεδρε. Η Αιθιοπία καταλαμβάνει ένα στρατηγικό πολιτικό και οικονομικό τμήμα της περιοχής και η Κομισιόν εξακολουθεί να υποστηρίζει την Αθιοπία με τα προγράμματα καταπολέμησης της Ένδιας και έχει σημειωθεί πρόοδος με την τοπική ασφάλεια και τις εντάσεις ε, που επηρεάζουν τις ιστορικές καταστάσεις των χωρών ιδιαίτερα στο κατέν, όπου η πρόσβαση στο κοινό παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένη. Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού. Μετά τις εκλογές του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την προετοιμασία των εκλογών του 2010, ιδιαίτερα στο συγκείμενο της πρόσφατα εγκριθής σας νομοθεσίας για τις ΜΚΟ και τις προσπάθειες του κ. Πυρτουκάν έξα. Η εσωτερική κατάσταση στην Ερυθρέα καθορίζεται εν μέρη από την συνοριακή διασυνοριακή αυτή διένεξη με την Αιθιοπία. Έχουμε σημαντικές ανησυχίες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την επισφαλή οικονομική κατάσταση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα, τα προγράμματα συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του κόσμου. Ο πολιτικός διάλογος που ξεκίνησε το 2008 αποτελεί μια καλή πλατφόρμα για την συνεχιζόμενη δέσμευσή μας και τη συνεργασία μας με τις αρχές της Ερυθρέας. Για να πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα, περιμένουμε να γίνει κάποια απτή πρόοδο στην Ερυθρέα. Όπως αναφέρετε και στο σχέδιο ψηφίσματός σας, η εικονική απομόνωση των ε, συνόρων μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας δεν θα οδηγήσει σε οριστική λύση αν δεν συνεδευτεί από κάποιο διάλογο για να ξομαλυθούν οι σχέσεις και η πρόσφατα η πρόσφατη διενέξη μεταξύ Ερυθρέας και Τσιμπούτη θα πρέπει να θεωρηθεί στο ευρύτερο συγκείμενο και θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να εξευρεθεί μια λύση από τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις διαδικασίες αυτές. Τώρα που τα στρατεύματα της Αιθιοπίας απομακρύνονται από τη Σομαλία, θα είναι σημαντική η συμβολή της Σομαλίας και της Ερυθρέας για την εξομάλυνση της κατάστασης. Για το Σουδάν, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την ανάλυση σας και με την ανάλυση των βουλευτών αναφορικά με την κατάσταση στο Σουδάν. Όντως, το 2009 θα αποτελέσει ένα έτος κλειδί, αν θέλετε, για το μέλλον της χώρας αυτής, για την ε, βία στον Ταρφούρ και τις δυσκολίες της, ε, του CPA, Όλα αυτά μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και όλη την περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε τους έντονους διαλόγους και να ασκήσουμε πίεση, να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση του Χαρτούμ για να συνεργαστεί απόλυτα και για το CPA αλλά και για το θέμα του Νταρφούρ. Οι αρχές αυτές, όπως και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς του Σουδάν, γνωρίζουν, γνωρίζουν πολύ καλά που είναι οι αρμοδιότητές τους και τι χρειάζεται να κάνουν στον Νταρφούρ θα πρέπει να λάβουν τέρμα η, στρατιωτική, η βία. Και θα πρέπει οι αρχές του Σουδάν να σέβονται τις αρχές τους και τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και τα δικαιώματα των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το CPA είναι απαραίτητο η κυβέρνηση του Χαρτούμ και του Σουδάν να ρυθμίσουν και να συμφωνήσουν για τις ε, διενέξεις τους, όπως είναι το πετρέλαιο, τα σύνορα, θέματα νομοθετικά και πολιτικά. Αν δεν γίνει αυτό, οι εκλογές του 2009 μπορεί να εξελιχθούν σε εκ νέου σειράξεις. Για τη Σομαλία τώρα, Πρόεδρε. Η ειρηνευτική διαδικασία στη Σομαλία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Η παρέτηση του Πρόεδρου Ιούσουφ και η απόσυρση του στρατού ανοίγουν μια νέα περίοδο αβεβαιότητας και κινδύνου, αλλά αποτελούν και μια ευκαιρία, αν θέλετε, για να ξεκινήσει μια συνεκτική πολιτική διαδικασία. Από πολιτικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί τις ε, ενεργειές της προς υποστήριξη της διαδικασίας του Τζιμπούτι, που θα πρέπει να οδηγήσουν στην εκλογή ενός ε, νέου Προέδρου και τον σχηματισμό ε, κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Δεν υπάρχει δεύτερο σχέδιο, αν θέλετε, για την διαδικασία της Τζιμπούτι. Αν δεν υπάρξει η περιφερειακή υποστήριξη που είναι απαραίτητη, η συμφωνία δεν θα έχει ουσιαστικά ε, ευκαιρίες επιβίωσης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η Κομισιόν υποστηρίζει και εξακολουθεί να υποστηρίζει τις σχετικές διαδικασίες. από όπου και να προέρχονται αυτές οι διεθνείς δυνάμεις, η εντολή τους θα πρέπει να εστιαστεί στην υποστήριξη της διαδικασίας του Τζιμπουτή και της σχετικής συμφωνίας. Έχουμε απαντήσει θετικά στο αίτημα για περαιτέρω χρηματοδότηση του Άμισον. Τέλος, Πρόεδρε, για το κέρος της Αφρικής εν γέννη, εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κέρας της Αφρικής η οποία βασίζεται στη στρατηγική του 2006 που υιοθετήθηκε με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα στην περιοχή αυτή μπορούν μόνο συνολικά να επιληθούν. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν σκοπεύει να προτείνει τον διορισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου για το κέρας. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το ΙΓΑΤ που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την πολιτική στην περιοχή. Μία δεύτερη συνεδρίαση για το Ίδωρ και για την ενέργεια και για τις συγκοινωνίες θα μπορούσε να αποτελέσει την έναρξη και θα προβλέπεται για το εγγύς μέλλον. Η συμμετοχή της Ερυθρέας που διαδραματίζει ένα ρόλο κλειδί είναι πραγματικά σημαντική για την επιτυχία, επιτυχία της στρατηγικής στο κέρας της Αφρικής. Ο Επίτροπος Μισελ και οι σχετικές πρωτοβουλίες τους έχουν ανοίξει προοπτικέ ω προ την κατεύθυνση αυτή και η γραμματεία του Ίγκατ έχετε σε επαφή με τις αρχές της Ερυθρέας για την μεταρρυθμίση και την αναζωγόνηση της Ίγκατ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μακρηγόρησα λίγο, αλλά τόσες χώρε βλέπετε τι να κάνουμε. Αν θέλουμε να πούμε δύο λόγια για όλες του παίρνει ώρα. Thank you very much. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν χρονικά όρια για την εισαγωγή μια συζήτηση ε, από πλευρά Συμβουλίου και Κομισιόν. Πρώτο αγοριστή, ο κύριο ε, Κάτσου Μάρεκ, θα μιλήσει εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο για δύο λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τις δηλώσεις που κάνετε σχετικά με το κέρδος ευρωπαϊκής. Η σημασία αυτής της περιοχής ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια Πρόκειται για προβλήματα διαθροτικού χαρακτήρα τα οποία ενισχύουν περαιτέρω άλλα προβλήματα στις γύρω περιοχές. Πρόσφατα συμμετείχα στην αντιστοπία του Κοινοβουλίου που μετέβη στην περιοχή και κατανόησα πόσο περίπλοκα είναι τα προβλήματα και πόσο ε, αλληλοσυνδέονται και αλληλοξαρτούνται οι χώρε αυτέ Το σχέδιο ψηφίσματος αναφερόμαστε σε σημαντικά προβλήματα όπως η περιφερειακή ασφάλεια, η επιστημική ασφάλεια, και όλα όσα αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει καμία εμβολία πως ε, βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της καταστάσεως είναι καλή βούληση και ο διάλογος ανάμεσα στους ηγέτες της περιοχής. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των ε, θεσμών στην περιοχή αυτή είναι κάτι το, το καλό, αλλά χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη συνεργασία με, τις, ε, με τα κράτη αυτά. δεν μπορούμε να κάνουμε έκκληση για διάλογο σε μια γειτονική χώρα αρνούμε παράλληλα τον διάλογο με μια άλλη χώρα της περιοχής. Αυτό δεν πρόκειται να έχει θετικά αποτελέσματα. Οι ηγέτες περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η άσκηση της εξουσίας ενέχει και ευθύνες. Αυτό το οποίο ζητάμε λοιπόν από τους ηγέτες του κέρατος της Αφρικής δεν είναι μόνο κάτι που είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές αρχές. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε οικουμενικές αρχές όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα απανταχού στη γη. Κανένα κράτος ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν ε, αρνηθεί αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η έννοια της ανάπτυξης μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Επ' δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σωστό μοντέλο προκειμένου να υπάρξει πρόοδο. Ευχαριστώ κυρία Αγκόμη για δύο λεπτά έχει το λόγο. Θα πρέπει να συναγάγουμε. Θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα και τις συνέπειες. Οι, οι χώρες γύρω από αυτή την περιοχή κατά το Κοινοβούλιο δεν ε, συμφωνηθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας. Υπάρχει το θέμα της δημοκρατίας, της καλής διακυβέρνησης και αυτό δεν το βλέπουμε. Θα πρέπει να μην εθελοτυφλούμε. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει κατάσταση του πληθυσμού. 29 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, είχαμε μια περίπτωση όπου είχαμε καταδίκη σε φυλάκιση διότι ζητήθηκε αμνηστία από την κυβέρνηση του Μελεσαναβή. Παραμένει στη φυλακή από το... με άλλους που είναι φυλακισμένοι από το 2005. Η Αιθιοπία επίσης έχει εγκρίνει νόμους σύμφωνα με το, σύμφωνα με τους νόμους ε, δημιουργούν ε, δυσκολίες όσον αφορά τις, μη κυβερνικούς οργανισμούς που είναι εκεί για να κάνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό που απαιτείται είναι να εφαρμόζονται και να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη Σομαλία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πληθυσμούς αυτής της χώρας και την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Επίσης, υπάρχει το πρόβλημα με την πειρατεία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν θα αποτελέσουν λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η, η, Ευρωπαϊκή, η Αφρικανική Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και να δώσουν λύσεις με δημοκρατικό τρόπο. Αλλά πραγματικά η κατάσταση δεν θα λυθεί και η κατάσταση είναι δραματική και το βλέπουμε και στο Σουδάν, στο Νταρφούρ, διότι μένουμε σε κενά λόγια, κενά λόγια από τη διεθνή κοινότητα και αυτό που χρειάζεται όμως είναι δράση. Και πραγματικά θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την κατάσταση της ατιμορρησίας των, των εγκληματιών. Συγγνώμη. Και έχουμε και την περίπτωση του διεθνού ε, Δικαστηρίου απέναντι από τον, ε, όσον αφορά τον πρόεδρο τη Ερυθρέα. Ο κ. Φανέκε, για ένα μισή λεπτό. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Το κέρα τη Αφρική είναι μια περιοχή όπου οι εσωτερικέ σειράξει εξακολουθούν να απονομεύουν την ασφάλεια και την ειρήνη προκαλούνται ανθρωπιστικές καταστροφές σε αυτή την σημαντικά στρατηγική περιοχή και κάθε πόλεμος τονίζει το ευάλωτο των κρατών αυτών. Στην καρδιά των πιο πολλών σειράξεων είναι η έλλειψη διακυβέρνησης δημοκρατικής και των ηγετών, το οποίο τόνισε σωστά η ομάδα του ΕΛΚ. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή αυτή είναι εκδημοκρατισμό, σεβασμό ε, του εθνικού και του διεθνούς δικαίου και πάνω απ' όλα εθνική συμφιλίωση. Για τη Σομαλία θα ήθελα να τονίσω ότι η παρέτηση του παρόν Πρόεδρου Γιούζεφ και η απόσυρση των ε, δυνάμεων, των στρατιωτικών δυνάμεων αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία και έχει έρθει η ώρα να μαζέψουμε τα κομμάτια για να πετύχουμε την ε, εσωτερική ειρήνη στη Σομαλία και θα πρέπει το Κοινοβούλιο της Σομαλίας να επιληφθεί της κατάστασης ειρηνευτικής διαδικασίας. Επίσης, αναφορικά με την ερηνευτική δύναμη στην Αφρική, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή εντολή. Όχι να φύγουν από το Μογκαντήσου οι δυνάμεις και να αφήσουν ένα κενό δυνάμεων. Υπάρχει όντως μια όθηση αυτή τη στιγμή στη Σομαλία, την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Η δύνα, αν θέλετε τα κενά δυνάμεων και ασφάλειας, θα πρέπει να πληρωθούν. Ιδάλλως θα παραμείνει η κατάσταση ως έχει στη Σομαλία. Ευχαριστώ από τους πράσινους. Ο κύριος Αμαζαγά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι το κέρας Αφρικής είναι μια περιοχή που μας ανισχύει ιδιαίτερα όχι μόνο για τη Σομαλία και το Σουδάν, αλλά και για τις τρεις χώρες οποίες ε, επισκεφθήκαμε προσφάτως ε, με τους συναδέλφους ε, Ερυθρέα, Τζιμπουτή και Αιθιοπία λοιπόν είναι τις αυτές χώρες οι οποίες γνωρίζουν την φτώχεια και επίσης παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα σε ό,τι φορά την φτώχεια είναι, έχουμε στοιχεία το ίδια οι δυσιαρχές της Αιθιοπίας θεωρούν ότι πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Ηνωμένο Έθνη ανεβάζουν αυτόν τον αριθμό σε 11 εκατομμύρια. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία τρομάζουν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης παραβιάζονται. Υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και στα τρία κράτη. Και θα πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε ιδιαίτερα την κατάστασή τους. Είναι πραγματικά παράλογο η σύγκρουση ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα. Υπάρχουν 250.000 στρατιώτες οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις σειράξεις και δεν θα ήθελα να κλείσω χωρίς να συγχαρώ την δράση του Επιτρόπου κ. Μισελ στην περιοχή προκειμένου να ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος. Ο πολιτικός διάλογος ο οποίος ε, θα πρέπει να συνεχιστεί, να αναπτυχθεί περαιτέρω, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ ε, αυστηροί σε ό,τι αφορά την ανθρώπινα δικαιώματα, ε, και ε, σταθερή σε ό,τι φορά τον σεβασμό τη δράση ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην περιοχή. Θα πρέπει να γνωρίσουμε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ ε, μεγάλο κύρο στην περιοχή. Επόμενο αγορητή του ονόματο τη Ενωρική Αριστερά, ο κύριος Πλούγκερ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το κέρας ε, της Αφρικής ξαναβρίσκεται πάλι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εκεί είναι σταθμεμένη η δύναμη Αταλάντη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δύναμη αυτή όπως και η Ρωσία και η ΕΠΑ και ο ΙΕ κάνει το εξής σφάλμα. Προσπαθεί με στρατιωτικά μέσα να ε, επιλύσει επιφανειακά τα προβλήματα. Και ο κύριος Κουσνέρ ε, πριν από δέκα δέκα χρόνια μετά το Σομαλό να δράσει με τον τρόπο αυτό. Το πρόβλημα είναι η άνεση κατανομή των πόρων, για παράδειγμα, και σε ό,τι αφορά την αλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει επίσης ουσιαστική κυβέρνηση και τα αιθιοπικά κατοχικά στρατεύματα έφυγαν από τη Σομαλία. Στο διάβο του σκότωσαν περίπου 200, σκοτώθηκαν 16.000 άνθρωποι. Στο Τζιμπουτί, για παράδειγμα, έχουν στρατιωτικές βάσεις σχεδόν όλες οι δυτικές ε, δυνάμεις, αλλά παράλληλα είναι αυταρχικό το καθεστώς. Ο κόσμος θα πρέπει να λάβει βοήθεια, όχι με τα μέσα, αλλά με ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλ Φον Δύο λεπτά. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η Σομαλία αποτελεί ένα κράτος ε, παρία με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό. Αναφέρεται αρκετά στοιχεία και η συνάδελφος Άννα Γκόμες ανέφερε θέματα τέτοια. Η πειρατεία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος, επειδή η πειρατεία αυτή είναι βαθιά ριζωμένη στην περιοχή αυτή και κατά δεύτερον πρόκειται για την προστασία των θαλάσσιων οδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δηλαδή συμφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της. Γι' αυτό υπάρχει, υπάρχει και αυτή η επιχείρηση Αταλάντη, που είναι η πρώτη τέτοια δραστηριότητα με βάση τη Μεγάλη Βρετανία και αυτό είναι καινούργιο στοιχείο. Και έχουμε και τον Άμαρχο Τζόνς που είναι υπεύθυνο, Βρετανός κι αυτός. Πρώτη εντολή της είναι να προστατεύσει την επιστηστική βοήθεια και να διασφαλίσει ότι όντω η επιστηστική αυτή βοήθεια καταφτάνει στη Σομαλία και κατά δεύτερον όμως και ο αγώνας η καταπολέμηση της πειρατείας. Είχαμε μια συζήτηση με την ηγεσία της επιχείρησης των Northwood και κατέστη σαφές ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία λείπουν ομολογουμένως, όπως για παράδειγμα ειδικά αεροσκάφη. Γιατί πρόκειται για την εποπτεία με περιοχή σε Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να επιδείξουμε ενδιαφέρον. Προκειμένου η Αταλάντη να επιτυξουμε ενδιαφερον επιτυχία. Αυτό είναι απαραίτητο αφενός για να προστατεύσουμε τις θελάσσιες οδούς μας, αλλά και αφετέρου για να συμβάλλουμε, έστω και με το μικρό αυτό το τρόπο, για την επίλυση του προβλήματος του αποτυχημένου κράτους της Σομαλίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσω τώρα το λόγο στον, στην κυρία Κρατού για 1,5 λεπτό. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τους συναδέλφους για ενημέρωση σε μια, όσον αφορά μια περιοχή η οποία είναι από τις πιο ε, επικίνδυνες στον κόσμο. Θεωρώ ότι στην Αφρική έχουμε τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Είχαμε το πρόβλημα της ξηρασίας στην Αιθιοπία, όπου εκατομμύρια κόσμου ε, πλήττονται από την πείνα ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε καλά. Είναι τραγικές αυτές οι περιοχές. Η κατάσταση ανθρωπιστική βρίσκεται είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε προβλήματα γενοκτονίας. Όλους αυτούς οι οποίοι διώκονται... Ε, το Τζιμπουτί, για παράδειγμα, είναι μια από τις πιο φτωχές περιοχές του, ε, του κόσμου. Γι' αυτό χαιρετίζω τους προλαλήσαντες. Έχουμε το κέρας Αφρικής όπου υπάρχει μια δύσκολη πολιτική και οικονομική ανάπτυξη και τα προβλήματα έχουν να κάνουν με προβλήματα διακυβέρνησης η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά θα πρέπει να υποστηρίξει αυτές τις χώρες στην ανάπτυξή τους και να μπορέσει να τις ενισχύσει ούτως ώστε να, τεθούν, να τεθεί τέρμα στις διενέξεις. Χρειάζεται ένας μεγαλύτερος διάλογος, έλεγχος όσον αφορά το εμπόριο όπλων και αυτά μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για το διάλογο και γι' αυτό θα πρέπει να ε, συμβάλλει περισσότερο να ενισχυθεί η, επέμβαση, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι χώρες θα πρέπει εκεί στην περιοχή να συμφωνήσουν, να πετύχουν μια συμφωνία όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, το 2001 είχαμε στην Ερυθρέα την περίπτωση του ενός Σουηδού υπήκοου, του Ίσακ, φυλακίστηκε και μετά από 7 χρόνια ακόμα δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του επίσημα. Για πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το ψήφισμα γίνεται μια μικρή αναφορά και δείχνει ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Ερυθρέα. Δεν είναι αποδεκτό, απαράδεκτο ένας δημοσιογράφος Ευρωπαίο υπήκο είναι φυλακισμένο, χωρί να υπάρχει κατηγορία εναντίον του. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία δέχεται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία μάλιστα έχει αυξηθεί τελευταία. Είναι καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και να ελέγξει τα θέματα τη βοήθεια. Τέρμα με τη διπλωματία τη σιωπηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχθεί όταν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα καταπαντούνται. Δημοσιογράφοι, ε, άτομα που είναι επικριτές της κυβέρνησης διώκονται και ε, καταπιέζεται ο λαός και πεινά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμα συζητεί ο Ντάβιτ Ίσακ και άλλους που είναι φυλακισμένοι στην Ερυθρέα να απελευθερωθούν. Αυτό θα ήταν ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να το απαιτήσουν είναι καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει στη δράση και να ε, επιβάλλει κυρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω και ο συνάδελφο μου από την ομάδα μου να ζητήσω την απελευθέρωση του Ντάβιτ Ίσακ. Επτά χρόνια ο Σιδός υπήκο Ντάβιτ Ίσακ είναι, υπήρξε φυλακισμένο χωρί δίκη κάτω από φοβερές συνθήκες σε μια δικτατορία. Χαίρομαι που έχουμε επιτέλους ένα κείμενο που ζητά την άμεση απελευθέρωση του. Ζητούμε αμέσως την απελευθέρωση του Ντάβιτ Ίσακ καθώς και άλλων φυλακισμένων δημοσιογράφων. Τι γίνεται, δεν έχει γίνει καμία δίκη και ποιο είναι το αδίκημα που έχουν κάνει. Το, αυτό που κάνανε ήταν έργο για τη δημοκρατία η βοήθεια προς την Ερυθρέα θα πρέπει να συνδυαστεί με μια, ένα αίτημα αποφυλάξης του Ίσα και άλλων φυλακισμένων δημοσιογράφων. Επίσης κυρώσεις να τεθούν και μεγάλες απαιτήσει από την Ευρώπη είναι κάτι το οποίο απαιτείται για να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση η, Ευρω... η Σουηδική κυβέρνηση είχε δράσει με αυτό που λέμε σιωπηλή ε, διπλωματία, αλλά μετά από 7 χρόνια νομίζω είναι καιρό για δράση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Στάνοκ. Ε, πρόεδρε, το κέρα τη Αφρική είναι ουσιαστικά μια τεράστια καταστροφή μετά από δεκαετίε ε, πείνα, περιβαλλοντικών καταστροφών, πολέμων, κακοδιαχείριση, πολιτική καταπίεση τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται καθημερινά και επίσης η κατάσταση φαίνεται ότι μπορεί να χειροτερεύσει και περαιτέρω. Οι διενέξεις μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας μπορούν να αναφλέξουν την κρίση να πάσα στιγμή. Η Σομαλία εξακολουθεί να πλήττεται από Ισλαμικό εξτρεμισμό που θα χειροτερεύσει αν η Αιθιοπία αποσύρει τα στρατεύματά της και μετά την απόσυρση, την παράτηση του Προέδρου η επιδημία της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας αναφέρθηκε. Πάντα υπάρχει φυσικά ο πειρασμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει τη θετική επέμβαση ως πανάκια, αλλά οι εμπειρίες του παρελθόντος καταδεικνύουν ότι αυτό ήταν τεράστιο σφάλμα. Ο Μπιλ Κλίντον έστειλε στρατεύματα στη Σομαλία, αλλά και αυτό εξελίχθηκε σε καταστροφή. Το μοναδικός λόγος αισιοδοξία είναι στην Σομαλία, πρώην ε, Βρετανικό protektorato. που ξαναπέκτησε την εξαρτησία του 1991. Έκτοτε η κυβέρνηση ήταν αρκετά ε, καλή και τα μέτρα ήταν αρκετά σοβαρά. Προσωπικά, όχι εκ μέρου της ομάδας μου. Ίσως είναι καιρός η διεθνής κοινότητα με την ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης να εξετάσει πιο σοβαρά την ε, αίτηση για την ανεξαρτησία της Σομαλίας. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια δύναμη σταθερότητας ε, στην περιοχή, στο χάος που επικρατεί στην περιοχή. Γιατί σίγουρα ο κόσμος της Σομαλίας ε, θα αναρωτιέται γιατί δεν αναγνωρίζουμε την de facto ανεξαρτησία τη περιοχή αυτή, αλλά την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Να περάσουμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye, λέει ο πρόεδρο. Πέντε ομιλητέ, ο κ. Νικολαύσκου πρώτα. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are într-adevăr toate motivele de a fi îngrijorată de situația creată în Somalia ανησυχούμε όσον αφορά την κατάσταση στη Σομαλία. Υπάρχει κενό εξουσίας και ίσως ε, λάθος άνθρωποι να καλύψουν αυτό το κενό. το ρόλο της ε, Αφρικανικής Ένωσης είναι το έργο της Αφρικανικής Ένωσης θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να δούμε το θέμα το, του ελέγχου στη θάλασσα περιπολίας. Αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά αν αυτό είναι η λύση. Είναι σαν να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μια αρρώστια χωρίς να ξέρουμε την αιτία της. Θα πρέπει η δράση σε διεθνέ επίπεδο να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία και σταθεροποίηση σε όλη την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές ευθύνες τόσο στη Σομαλία όσο και σε όλη την Αφρικανική ε, περιφέρεια. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για πολλούς λόγους. Όλο και πιο πολύ αυξάνονται οι πειρατείες σε αυτή την περιοχή έξω από τη Σομαλία και αυτό έχει επιπτώσει στην ε, διακίνηση, την ε, εμπορική που γίνεται στην περιοχή και διαπιστώνουμε ότι αυτά σε ομάδες που δρούν εκεί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ε, προηγμένη τεχνολογία και ελέγχουν τις ακτές. Στη Σομαλία δεν υπάρχει κεντρική κυβέρνηση ικανή να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα. Η διεθνής κοινότητα έχει μια ευθύνη όμως εδώ. Η πειρατεία, όποια και αν είναι αυτή, με οποιοδήποτε συνθήκες και αν γίνεται, είναι δραστηριότητα η οποία εναντιώνεται στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό που, μπορεί να κάνει, ε, που κάνει η διεθνή κοινότητα στην περιοχή ε, δεν είναι αρκετό για να ανθρωπίσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκλώθηκε ο κατάλογος των αγορητών. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Να αναφερθώ πρώτα στις παρατηρήσεις που έγιναν και να συναγάγω κάποια συμπεράσματα. Ο Λε Σμιτ, Εύα Σβένσον αναφέρθηκαν στον δημοσιογράφο David Ιζακ. Προσπαθούμε να πετύχουμε την απελευθέρωσή του. Η κυρία Άννα Μαρία Γκόμες αναφέρθηκε στον κύριο Μπέρτουκαν το Συμβούλιο γνωρίζει πολύ καλά την υπόθεση Μπερτουκάν. Πρόκειται για μια περίπτωση, μάλλον πρόκειται για κάποιον που συνελήφθη το 2005 συνάδελφος αναφέρθηκε στην περίπτωση αυτή και Πράγματι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει δράση για την απελευθέρωσή του. Και τώρα να κάνω πέντε παρατηρήσεις. Να σας πω πρώτα απ' όλα πως ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η αντιπροσωπεία σας ε, που μετέβη στην ε, περιοχή. Επίσης με ο κύριο και ο κύριο Χάτσκινσον να σας διαβεβαιώσω πως ε, υπό τσεχική προεδρία θα υπάρξει μια συνέχεια του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή που αποφάσισαν οι προκατοχοί μας ε, με αποτελεσματικό τρόπο. Θα φροντίσουμε να περιορίσουμε την ε, πειρατεία και εκτιμάμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Γαλλικής Προεδρίας που προώθησε την ανάπτυξη της ε, πρώτης ε, ναυτικής δύναμης ε, στην περιοχή. Μια δεύτερη παρατήρηση. Η επιχείρηση Αταλάντη έχει ήδη προλάβει κάποιες πειρατείες, τις έχει αποτρέψει και μετά από μερικούς μήνες λειτουργίας της βλέπουμε αυτά αποτελέσματα. Η Αταλάντη φυσικά είναι ένα μέτρο βραχυπρόθεσμο, αλλά ήταν απαραίτητο μέτρο για να καταπολεμήσουμε την πειρατεία. Θα φροντίσουμε να βρούμε μια μακροχρόνια λύση του προβλήματος της Σουμαλίας στο Συμβούλιο, υποστήριζε τη δικασία του Τζιμπουτή για την ε, μεταβατική κυβέρνηση και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο Β αναδίπλωσης. Η Σομαλία είναι σημαντικό τμήμα για την διαδικασία του Τζιμπουτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως συνεχίζει να στηρίζει την Αφρικανική Αποστολή Άμισον στην Σομαλία. 20 εκατομμύρια ευρώ έχουν χορηγηθεί για την περίοδο Δεκέμβρη 2008 και Μάη 2009. Τέταρτον, τις ε, άμεσες επαφές που προβλέπουμε για την επανάληψη του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις αρχές ε, της περιοχής σε υπουργικό επίπεδο βλέπουμε πως οι ειρηνευτικές ε, συνομιλίες στην Σομελία απέδωσαν. Οι αρχές λοιπόν ε, μπορεί να αποτελέσουν έναν εταίρο κλειδί προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Σομαλία. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αφορά το θέμα μιας μεγαλύτερης δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά την αθεώρηση της στρατηγικής για το κέρας Αφρικής ε, της η, Αφρική, η Κομισιόν είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας και αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με την συνέχεια της πολιτικής μας στην περιοχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να κάνω λίγα σχόλια για την σύντομη αλλά πολύ σημαντική αυτή συζήτηση. Καταρχάς για τη Σομαλία. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα όλα αυτά τα σχόλιά σας, όλες αυτές τις προτάσεις και με ενθαρρύνει το γεγονός ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης αλλά και για τις δράσεις που θα πρέπει να αναλευθούν. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε όντω το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και τους βασικούς, αν θέλετε, παράγοντες του Ισλαμικού κόσμου για να εξευρεθεί μια βιώσιμη πολιτική λύση στη Σομαλία προκειμένου να τελειώσει επιτέλους ε, η καταστροφή αυτή. Η Κομισιόν στο τομέα αυτό θα παρέχει πολιτική αλλά και οικονομική ενίσχυση για τη διαδικασία του Τζιμπουτή. Συμφωνώ με την κυρία Γκομές ότι οι χώρες του κέρατος όντως αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Μας ανησυχούν αυτές οι τεράστιες αυτές προκλήσεις, αλλά φοβούμαστε ότι σε σχέση με το άρθρο 9 της Συμφωνίας του Κοτονού είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην καλή διακυβέρνηση και στα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, με τον πολιτικό διάλογο και με σαφή οριοθέτηση για την ε, επισητιστική ασφάλεια. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μία από τις προτεραιότητες του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου και στο πλαίσιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πέρα από το φάκελο του EDF υπάρχει πλέον, υπάρχουν και άλλα κονδύλια στο μέσο Food Facilities, 100 εκατομμύρια ευρώ από το 2009 στο 2011. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι συνειδητοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση του Σουηδού πολίτη Ιζακ, της ε, πολίτη Ιζακ, που βρίσκεται ακόμα υποκράτησε ο συνάδελφος μου Λίς Μισελ έχει μιλήσει στον πρόεδρο Ισάγια στην τελευταία επίσκεψή του τον Ιούνιο του 2008 και συνεχίζονται τα διπλωματικά παρασκήνια για το θέμα αυτό. Φυσικά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνουμε δεσμευμένοι για την επίλυση της ανθρωπιστικής κατάστασης και στην Ερυθρέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έτσι κλείνει η συζήτησή μας αυτή. Να σας ενημερώσω ότι έλαβα κοινό σχέδιο ψηφίσματος από έξι πολιτικές ομάδες, ΕΛΚ, ΑΛΔΕ, Σοσιαλιστές, Πράσινοι και η UEN αλλά και η GUE NGL. Ε, ε, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξής μας, το οποίο είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας. Ο συνήθως θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Κύριε Υφυπουργέ Βόντρα, έχετε το λόγο.